Πρέπει να σκοτώσουμε ένα σοσιαλιστή. Εντάξει. Ευχαριστώ. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ακολουθούμε επίση με την αντίρρηση βάσει του άρθρου 106 έγκριση γενετικά τροποποιημένου αραβοσιτού νίκαιη 603 επιτάφη 25. Ο εισηγητής είναι ο Μπάτς Θάες. Λοιπόν, πρέπει να ψηφίσουμε τα στοιχεία 13 και 14 γιατί αφορούν το ίδιο αντικείμενο. Στο 14 είναι η συγγήτρια Σιλβί Γκοντίν το άλλο θέμα. Εάν δεν γίνει δεκτό. Ψήφισμα Σιλβί Γκοντίν άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε το σχέδιο του Bart Stiles και άλλων. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Εντάξει. Πέρας. Εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στο σημείο 15, την έκθεση Childers, για τη λογοδοσία, την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Νέσσα Childers είναι η Αρχίζουμε να ψηφίσουμε με την συμβαστική τροπολογία 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά. <clears throat> Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 6. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 <clears throat> υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 ψήφι υπέρ κατά αποχές έλεγχος. The vote is closed. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορριφθήκε 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 21 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά <clears throat> αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 23 υπέρ. Κατά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 <coughs> Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος για το δεύτερο τμήμα τη 24. Ψηφίσατε όλοι και όλες. Πέρας. Απορρίπτεται. 47 με προφορική τροποποίηση από την ομάδα ECR. Έχετε αντίληψη για την προφορική τροποποίηση? Όχι. Όχι. Έχετε? Όχι, δεν έχετε. Λοιπόν, ψηφίζουμε την 47 με την προφορική τροποποίηση. Υπέρ. Κατά. Αποχές συγκρίνεται. 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 υπέρ κατά έλεγχος για την 59 ψήφισατε όλοι πέρας εγκρίθηκε. 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ κατά αποχές κάνουμε έλεγχο. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 52. <clears throat> Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 53. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 54 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές έλεγχος Και το δεύτερο τμήμα της 54. Όλοι ψηφίσατε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 55 πάλι σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Το δεύτερο τμήμα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έλεγχος για την 63 μάλιστα ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίθηκε 64 σε 3 τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 67. Ψήφι υπέρ. Κατά Αποχές εγκρίνεται. Το σχέδιο γνωμοδότησης όπως έχει τροποποιηθεί ηλεκτρονικά. Άρχεται. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Όμορφο να δεκτώ. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια, την κυρία Τσίλντες. Can I ask to all uh, the members and other people who are... Να ζητήσω από όλους όσοι δεν ενδιαφέρονται για το επόμενο σημείο να εγκαταλείψουν την αίθουσα ησύχως. I ask another time to all the people who are not interested in the next. Επαναλαμβάνω λοιπόν όσοι δεν ενδιαφέρονται για το επόμενο σημείο της μισής διατάξεως να εγκαταλείψουν την αίθουσα. Πρόκειται για το σημείο 16. Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για τον Συντονισμό των Οικονομικών Πολιτικών. Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 2016 και θα ήθελα να δώσω αμέσως το λόγο στον εισηγητή Αντρέη Κόβατσεκ. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα προσπαθήσω συντομία να εξηγήσω τα βασικά σημεία που με απασχόλησαν με αυτήν την γνωμοδότηση. Όπω γνωρίζετε, Για αυτή η ετήσια επισκόπηση που αφορά στον, το, το 2016 δημοσίευσε και πριν από μερικού ε, μέρε. Και θέλει να εξετάσει και να προωθήσει την ανάπτυξη σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς η ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια ήταν πολύ χαμηλή. Έχει ιδιαίτερη σημασία να επαναλάβουμε την πρότασή μας να, ε, και να καταδείξουμε στους πολίτες μας ότι έχουμε μια ε, στεναρή στρατηγική που όχι μόνο θα ε, επιταχύνει την ανάκαμψη αλλά θα προχωρήσει σε μια ε, βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Η στρατηγική του 2020 δεν έχασε την σημασία της και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πλαίσιο για την πρόθεση της απασχόλησης και της ανάπτυξης. Ε, να διορθωθούν τα σφάλματα της στρατηγικής αγώνας. Να υπάρξει λοιπόν μια στρατηγική η οποία τώρα στα μέσα του κύκλου θα πρέπει να ε, επαναπροωθηθεί. Η ανάπτυξη έχει αρχίσει να επανέρχεται και οι συνθήκε είναι, καλέ είναι καλές για να στοχεύσουμε σε μια μακροπρόθεσμη ανάπτυξη για την Ευρώπη. Η, στρατηγική, η αναφερμένη στρατηγική του 2020 έχει συμπεριληφθεί καλύτερα στην διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξάμεινου για την παρακολούθηση της ε, ανάπτυξης και των εξελίξεων περιβαλλοντικές ε, και κοινωνικέ πτυχέ θα πρέπει να δραματίσουν σημαντικό ρόλο στον εξάμεινο αυτό, διότι οι προποθέσει για ανάπτυξη είναι σημαντικέ σε αυτούς τους τομείς. Συμφωνούμε με την νέα προσέγγιση της Κομισιόν για την στόχευση σε στόχους κλειδί, για, ειδικά για την πράσινη ανάπτυξη και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, τη βελτίωση της ε, ε, ασφάλεια ε, των εφοδιασμού. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι αποτελεί το κλειδί για την πρόθεση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων ε, περιβαλλοντική και, και τα θέματα, περιβαλλοντικά προβλήματα και τα θέματα υγείας συμβάλλουν για την εφαρμογή της πολιτικής αυτής, στρατηγικής αυτής συγγνώμη, για το 2020 οι αριθμοί καταδεικνύουν ότι ακόμα και κατά τα χρόνια της ύφεση η απασχόληση σε αυτούς τους τομείς ε, αναπτύχθηκε. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε ότι η κάλυψη των περιβαλλοντικών και των και των πτυχών υγείας ε, τα τελευταία χρόνια μειώθηκαν σημαντικά από 41 συστάσεις το 2014 σε 14 το 2015. Πάντω είναι συγκαριστή σαφέ ότι αυτό δεν οφείλεται σε μια ανεπαρκή πρόοδο τους ε, λογοτομείς. Η εφαρμογή αυτών των συστάσεων συχνά δεν προωθήθηκε διότι ήταν ασαφής ή στόχευσε μόνο σε θέματα περιβαλλοντικά και ε, ε, θέματα δημοσιονομικά. Θα πρέπει να στην Κομισιόν να προωθήσει την ε, σύγκληση ε, των οικονομικών δικτών. Οικονομικών δικτών. Αυτός θα ήταν ένας κατάλληλος τρόπος για να αρχίσουμε ε, να αποτρέψουμε τα, τα κράτη-μέλη ώστε να περιορίσουν τις δαπάνες και να μην λαμβάνουν υπόψη τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Θα πρέπει να δώσουμε σταθερή βάση για το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς επίσης και το, να τονίσουμε και το ζήτημα της κυκλικής οικονομίας. Επίσης να πω μερικά λόγια για το ότι πιστεύω ότι η, η υγεία θα πρέπει να αποτελέσει ένα σημαντικό τμήμα και να της αποδοθεί ιδιαίτερη σημασία. Η πραγματικότητα μας δείχνει ότι η καλύτερη συνεργασία απαιτείται και στον τομέα αυτό για να μπορέσουμε να συμβάλλουμε ιδιαίτερα στον τομέα της ε, ανάπτυξης των θέσεων και υψηλής ποιότητας απαιτείται να μειωθεί η διαφορά σε αυτούς τους τομείς. Θα ήθελα να σταματήσω το σημείο αυτό και να ακούσω τους ε, συναδέλφους μου όπως τον Σκιώδη Συγητή σε αυτό το θέμα και να τους ευχαριστήσω ε, Ευχαριστώ. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τώρα με το στοιχείο ηγητές, ξεκινώντας από τον κύριο Τζουρίγκο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή για την εργασία του και θέλω να εστιάσω την παρέμβασή μου σε τρία σημεία για την ε, ανακοίνωση της Κομισιόν, για την έκθεση του εισηγητή και για την συνέχεια πρέπει να δώσουμε. Η ανακοίνωση της Κομισιόν τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο πρέπει να συνδυάζει τα οικονομικά θέματα με τα κοινωνικά και τα περιβαλλοντικά θέματα. Αυτό όμως δεν έχει γίνει. Εμείς βλέπουμε αυτή τη στιγμή σε μία ε, ανάγκη να έχουμε μία σύγκληση η οποία να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες για επενδύσεις, για κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. <clears throat> Θα ήταν πολύ θετικό λοιπόν να συμπεριλάβουμε στο έγγραφο αυτό για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο τις προκλήσεις που χρειάζονται να αντιμετωπιστούν. χάρη τις προτάσεις μας για την ψηφιακή, ψηφιακό θεμετολόγιο, για την ενεργειακή μετάβαση, τους στόχους της Ευρώπης 2020 που θα πρέπει και αυτοί να αναφερθούν όπως λέει και ο εισηγητής μου. Ο εισηγητή εστιάζει στα ουσιαστικά θέματα στην ενσωμάτωση στρατηγική Ευρώπη 2020 στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Τονίζει τη σημασία τη κυκλική οικονομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη ενέργεια και την ανάγκη να έχουμε μια συνολική προσέγγιση στα θέματα υγεία. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι ακόμα. Ξέρω ότι είναι περιορισμένο σε αριθμό λέξεων, αλλά μπορούμε να πούμε περισσότερα. Έχουμε ενώπιόν μας και τη διάσκεψη για το COP21 για την κλιματική αλλαγή, τα θέματα αντιμετώπισης του ρεύματος των ε, προσφύγων. Θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη έμφαση στα θέματα του περιβάλλοντος και της υγείας μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Οι στόχοι της Ευρώπης 2020 θα πρέπει να ενσωματωθούν, η ευφυής και περιεκτική δηλαδή και βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτές οι ε, δεσμεύσεις θα πρέπει να οδηγήσουν σε θέσεις εργασία ποιότητος γιατί η βιωσιμότητα δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται αντιμέτωπο, αλλά υπέρ της δημιουργίας θέσεων εργασίας ποιότητας μπορούμε να τονίσουμε επίσης την ανάγκη να υπάρχει μεταλαμβάνευση των πρακτικών στον τομέα της υγείας και επίσης μέσα στα έγγραφα αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και το μέλλον επέκεινα του 2020 και τις δεσμεύσεις που πρέπει να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε τομείς όπως η υγεία να σκεφτούμε λοιπόν πώς θα μπορέσουμε να σχεδιάσουμε την μελλοντική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις δεσμεύσεις που θα πρέπει να αναλάβουμε. Πασφυρτός έχουμε μια πολύ καλή βάση εκκίνησης σε αυτή τη γνωμοδότηση. Επομένως δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ τη βασική ιδέα που είναι ότι πρέπει στο έγγραφο του Ευρωπαϊκού Εξάμεινου θα πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο η πολιτική του προϋπολογισμού και η πολιτική της βιώσιμης ε, ανάπτυξης και της απασχόλησης. Ευχαριστώ. Ο κύριο Φαρία. Ehm, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή, τον κύριο Κόβατσεφ και να τον ευχαριστήσω για την πολύ καλή εργασία που έχει παρουσιάσει με την, με την έκθεσή του, με την γνωμοδότηση αυτή της Επιτροπής ΕΝΒΗ σε σχέση με την ε, ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι αυτά που λέει είναι αρκετά πλήρη και συμφωνώ γενικά με τα σημεία τα οποία έχει εξάρει ο εισηγητής. Νομίζω ότι η αποδοτικότητα στη χρήση των πόρων και μια μεγαλύτερη έμφαση στην πράσινη ανάπτυξη μπορούν να οδηγήσουν την Ευρώπη σε μεγαλύτερη ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Σε ό,τι αφορά το αναλυτικό τμήμα της έκθεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις επενδύσεις, νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να προωθούμε συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να κάνουμε μια προσεκτική ανάλυση των εργαλείων που έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Ένωση και εγώ θα τονίζω τη σημασία του EFSI για τις στρατηγικές επενδύσεις. Οι επενδύσεις αυτές θα πρέπει να κατευθυνθούν με τον σωστό τρόπο, κυρίως στους τομείς όπου είναι δυνατό να υπάρξει μια μετάβαση προς μια βιώσιμη ανάπτυξη και που συνάδουν με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για το 2020 να προωθήσουμε την τεχνολογική καινοτομία στο, επίσης και στο ενεργειακό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα πρέπει να πιο ευφυές και καλύτερα διασυνδεδεμένο, όπως είπε και ο κύριος Ζωρίνιο, μόνο με τις τεχνολογίες αυτές μπορούμε να προχωρήσουμε πιο μια πιο βιώσιμη και αποδοτική οικονομία που θα έχει καλύτερη χρήση των σπανίων πόρων, φυσικών πόρων και που θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και μεγαλύτερη ε, δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Για το δεύτερο πυλώνα αυτής της ανάλυσης, το θέμα της ε, ανάπτυξης, ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη δομικές παραμέτρους όπως είναι η μορφή του σχολικού και εκπαιδευτικού γενικά συστήματος που θα επιτρέψουν μια καλύτερη προσαρμογή στην αγορά και καλύτερη προσαρμογή των ανθρωπίνων πόρων οι οποίοι θα πρέπει να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για να συμβάλλουν στο να υπάρξει μια οικονομία η οποία θα έχει μεγαλύτερη δυνατότητα ε, δημιουργίας προσθέμενης αξίας. Υπάρχει, καλύτερη, υπάρχει ανάγκη καλύτερης διασύνθεσης μεταξύ του συστήματος παιδείας με το σύστημα τεχνολογικής εκπαίδευσης, μάλλον καινοτομίας, και καλύτερης μετάβασης μέσα στο χώρο εργασίας από το σχολικό σύστημα. Θα πρέπει επίση να βελτιώσουμε και την αποτελεσματικότητα του συστήματο κοινωνική ασφάλεια και εδώ συμφωνώ απόλυτα με τον εισηγητή. Είναι απαραίτητο το σύστημα αυτό να είναι αποτελεσματικό αλλά να διατηρεί και την ποιότητα και τη βιωσιμότητά του. Και πιστεύω ότι δεν είναι μονάχα αυτός ένα σημαντικός τομέας ε, δραστηριότητας, αλλά και μία πηγή απασχόλησης και εδώ είναι μία από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο που την εκτιμούν ιδιαίτερα οι πολίτε. Πρέπει επίση να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την καλύτερη πρόσβασιμότητα των υπηρεσιών υγειονομική περίθαλψη και θα ήθελα επίση να τονίσω ότι, όπως αναφέρει ο εισηγητής βέβαια, τονίζει ότι ο συγητής, ότι ο τομέας της υγείας θα πρέπει να ε, αντιμετωπιστεί λίγο περισσότερο και να δοθούν περισσότερες επενδύσεις στον τομέα αυτό. <clears throat> σε ό,τι αφορά τι δημοσιονομικέ πολιτικέ, έχουμε ακόμα τρόμο να διατρέξουμε φυσικά για να μπορέσουν αυτές να οδηγούν σε βιώσιμη ανάπτυξη και να προωθούν τι επενδύσει. Θα πρέπει να βρούμε μηχανισμούς ε, δημοσιονομική αντιστάθμιση σε ό,τι αφορά τεχνολογική καινοτομία και την προστασία του περιβάλλοντος και συγχρόνως με τον τρόπο αυτό να μπορέσουμε να προωθήσουμε την λεγόμενη κυκλική οικονομία. Και τελικά η διαδικασία εφαρμογής του κύκλου του εξαμήνου θα πρέπει να βελτιωθεί, θα πρέπει να υπάρξει και μεγαλύτερη συμμετοχή και των εργαζομένων στη χάραξη στρατηγικών για την απασχόληση και επίση αντιμετώπιση τη σχολική αποτυχία και του κοινωνικού αποκλεισμού να τονίσουμε ότι πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μας τη βιώσιμη ανάπτυξη, να έχουμε στρατηγικές βιώσιμες σε εθνικό επίπεδο και να κινηθούμε προς μια μεγαλύτερη εσωτερική σύγκληση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά την υποστήριξη προς τους που και εδώ θέλω να τονίσω αυτά που είπε ο κ. Ζωρίνιο, είναι απαραίτητο να αναφερθούν και αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε κ. Σλέκ τώρα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Θα συνεχίσω στα κροατικά. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κόρατσεφ γιατί πάντα επιστρέφουμε στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Στηρίζω λοιπόν όλα όσα προτείνονται εδώ. Θα τονίσω διάφορα στοιχεία όσον αφορά την κυκλική οικονομία. Αυτό πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και η νομοθεσία για την διαχείριση των αποβλήτων. Στηρίζω επίσης τη μείωση της εξάρτησης από την ενέργεια και στηρίζω και τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Πρέπει πράγματι να στηρίξουμε τα θέματα αυτά. Όσον αφορά τώρα την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, πρέπει να εκτιμήσουμε μέσα σε όλα και το θέμα των κλιματικών αλλαγών. Οι μεταρρυθμίσεις δευθυντικές ε, και άλλες πρέπει να συνάδουν με μια τέτοια πολιτική. Η κοινωνία των πολιτών πρέπει να έχει μια περισσότερο δυνατή φωνή. Υπογραμμίζω επίσης ότι δεν τονίζεται αρκετά αυτό το τελευταίο στοιχείο και οι χώρες μέλη θα πρέπει να στηρίξουν και τα εκπαιδευτικά συστήματα. για να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης, πράσινες θέσεις απασχόλησης, και σε αυτό θα βοηθήσει σίγουρα η Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ωραία, ποιος άλλος θέλει το λόγο. Δεν βλέπω. Κανένα, ο κύριος Κοντέσκου, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τώρα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον που δείχνετε στο θέμα αυτό του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ευχαριστώ και τον εισηγητή σας. Υποδεχόμαστε με ικανοποίηση την προσπάθεια αυτή. Στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και εμείς συνεργαζόμαστε και με την Γενική Διεύθυνση ΦΙΝ και τα τελευταία χρόνια είναι αλήθεια ότι επικεντρωνόμαστε περισσότερο στην μακροοικονομική σταθερότητα και διάφορους λόγους. Η Επιτροπή θέλει καλύτερη εφαρμογή των συστάσεων κλπ. Τελευταία, όπως σας είπα, συνεργαζόμαστε στενά. Έχουμε στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι η περιβαλλοντική πολιτική μπορεί να βοηθήσει την οικονομία και την απασχόληση. Άρα να έχει θετικές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας. Οι κεντρικές υπηρεσίες δουλεύουν πάνω σε αυτό. Και τώρα, την περίοδο 2015-2016, θα θέλαμε το περιβάλλον να περιλαμβάνεται στις αναχώρα εκθέσεις, ακόμα και αν δεν είναι οι ίδιες οι χώρες που το αναφέρουν. Για τις χώρες μέλες έχουμε μία ομάδα εμπειρογνωμόνων που κοιτάει πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου στο περιβάλλον. Πρόεδρος. Ο εισηγητής και πάλι για να κλείσουμε τη συζήτηση. Παρακαλώ κύριε Κόβατσεφ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους συναδέρφους για τα σχόλιά τους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλα όσα τονίζετε είναι σημαντικά και πιστεύω ότι μαζί θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια καλή έκθεση, σε ε, καλές συστάσεις όσον αφορά το περιβάλλον, την εξοικονόμηση ενέργειας, την εκπαίδευση, τις δεξιοτεχνίες γύρω από την ενέργεια και το περιβάλλον για πράσινες θέσεις απασχόλησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι έχει στοιχεία που δείχνουν ακριβώς ότι οι θέσεις απασχόλησης σχετικές με το περιβάλλον μπορούν να γεννήσουν ακόμα περισσότερες θέσεις εργασίας. Τα θέματα υγείας ίσως να μην λαμβάνονται παρκώς υπόψη. Στόχος κάποιων χωρών για τα θέματα υγείας είναι να αποφύγουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει συστάσεις σε αυτό το τομέα και επικαλούνται την επικουρικότητα. Εγώ όμως πιστεύω και σας ζητάω να το στηρίξετε κι εσείς ότι χρειάζεται μια πιο ισχυρή διάσταση της υγείας μέσα στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι και προσβλέπω σε καλή συνεργασία με τους σκιώδεις εισηγητές. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Τώρα πρέπει να διακόψουμε για λίγο. Περιμένουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας έρθει για το επόμενο θέμα. Η προθεσμία είναι η 8η Δεκεμβρίου. Στα αγγλικά προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Γιατί πάντα έχουμε το πρόβλημα χρόνου. Θα έχουμε έκτατη συνεδρίαση στις 21 Ιανουαρίου στο Στρασβούργο και στην ΕΚΟΝ ψηφίζει, η ΕΚΟΝ ψηφίζει το Φεβρουάριο και θα πάει το θέμα στην Ολομέλεια το Μάρτιο. Αυτά λοιπόν, διακοπή λίγα λεπτά μέχρι να έρθουν οι εκπρόσωποι της Επιτροπής. o'clock. Η ώρα είναι πέντε. Ας ξεκινήσουμε. Έχουμε το ζήτημα σχετικά με την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας θα δώσουμε το λόγο στην Κομισιόν, την οποία και ευχαριστούμε που παρίσταται. Ξεκινήσουμε από μία ερώτηση του Σεπντάνς και δίνω το λόγο στην Κομισιόν για τις απαντήσεις. Την Κομισιόν έχουμε την κυρία Βέντινγκ. Και να ξεκινήσουμε με την πρώτη απάντηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Ε, για την πρώτη ερώτηση, η ερώτησή μας έχει εξή. Η Κομισιόν δεν έχει δει τα τελευταία προγράμματα της Βρετανικής Κυβέρνησης για την ποιότητα του αέρα σχετικά με την εφαρμογή περί ποιότητας περί αέρα Ζητήσαμε για μια περαιτέρω ενημέρωση και αυτή μα χορηγήθηκε από τι αρχέ του Ηνωμένου Βασιλείου. Γνωρίζετε ότι τα προγράμματα ολοκληρώνονται στα τέλη του έτου και περιμένουμε την τελεκτή εκδοχή τη βρετανική κυβέρνηση περί ποιότητα του αέρα και δεν μπορούμε προς το παρόν να επιβεβαιώσουμε ότι τα προγράμματα θα μα διασφαλίσουν την συμμόρφωση. Καταλαβαίνουμε ότι τα προγράμματα καλύπτουν 38 ζώνες και υπάρχουν σημαντικές διαφοροποίησεις σε αυτές τις περιοχές. για σε της Κομισιόν περιμένει ότι θα εφαρμοστούν φιλόδοξα μέτρα μετά από την ανακοίνωση αυτού του προγράμματος. Επίσης καταλαβαίνουμε ότι το πρόγραμμα αυτό συμμορφώνεται ε, ε, ώρες της ζώνης το 2020 υπάρχει και μια προθεσμία καταληκτική το 2025 σε εθνικό επίπεδο ο ακρογωνίος λήθος της προσέγγισης ε, φαίνεται ότι αποτελεί ένα νέο εργαλείο όπως επίσης και εντατικοποιημένες προσπάθειες αναφορικά με τον εξηλεκτρισμό του του, των οχημάτων. Οι ρήποι στον αέρα, του αέρα μάλλον δεν έχουν ακόμα υπολογιστεί και ποσοτικοποιηθεί. Τα τελικά προγράμματα που σας είπα θα υποληθούν έως τα τέλη του έτους. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα που να μου επιτρέπει να σας πω περισσότερα για το πρόγραμμα που θα ισχύει σε από το 2025, 15 χρόνια λοιπόν από την αρχική εφαρμογή του προγράμματος. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ. Κύριε Γκλώδο, θέλετε να πείτε κάτι. Ε, ich glaube, dass schon viele Dinge Νομίζω ότι έχουν ήδη ε, λεχθεί όπως αναφέρθηκε από την Κομισιόν η επικαιροποίησή της θα βοηθήσει να προχωρήσουν τα πράγματα και μέχρι το τέλος του χρόνου περιμένουμε μια πιο οριστική πρόταση ώστε να δούμε κατά πόσο μπορεί να κινηθεί μια διαδικασία για παραβίαση των συνδικών συγκεκριμένα του άρθρου 23. Οπότε από αυτή την άποψη νομίζω ότι έχει λυθεί το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στον κύριο Πετιτσίνη. Μήπως μπορείτε να απαντήσετε το ερώτημα του κυρίου Πετριτσίνη για την μη συμμόρφωση και τις διαδικασίες επί παραβάση την τέταρτη ερώτηση συγκεκριμένα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να σας υπενθυμίσω ότι τα κράτη-μέλη έχουν την υποχρέωση να επιτύχουν την τήρηση των οριακών τιμών για την ποιότητα του αέρος όπως αναφέρεται στην ε, ε, οδηγία για την ποιότητα του αέρος, αλλά η οδηγία της δεσμεύει ως προς το στόχο και όχι ως προς τους τρόπους με τους οποίους θα επιτύχουν κάτι τέτοιο. Μέσω στα πλαίσια της εφαρμογής των κανόνων για τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κάτι έχουν και άλλους τρόπους για να μπορέσουν να επιτύχουν τους στόχους της νομοθεσίας για την ποιότητα της ατμόσφαιρας του αέρος. Οικονομικά εργαλεία ή επίσης αντιμετωπίζοντας εκπομπέ από ορισμένου τομεί εν ε, όψη των σημαντικών επιπτώσεων στην υγεία της ε, ρήπανσης του αέρος, η Κομισιόν θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για να εξασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας για τα θέματα αυτά. Η υπέρβαση των ε, ορίων για το διοξείδιο του αζότου που έχουν θεσπιστεί από την νομοθεσία του 2010 στον αστικό χώρο φυσικά οφείλονται στην χρήση αυτοκινήτων με κινητήρες δίζελ που όπως έχει επιβεβαιωθεί πρόσφατα φυσικά εκπέμπουν πολύ περισσότερο από ό,τι προβλεπόταν από το πρότυπο Euro 5 για το 2030 που είναι το πλαίσιο το οποίο έχει αντιμετωπιστεί στην πρόταση της Κομισιόν για την ε, τροποποίηση οδηγίας NEC... προβλέπεται να υπάρξει η εφαρμογή των τεστ σε πραγματικές συνθήκες και θα εξασφαλίσει ότι οι εκπομπές των ε, αυτοκίνητων diesel θα είναι πιο κοντά στην αρχική ανάλυση που διέτρεχε την επαναθεώρηση του ΝΕΚ. Παρακαλώ κύριε Ευχαριστώ πρόεδρε. Η ερώτησή μου και κυρίω κυρίως στο εξή. Οι υπολογισμοί των επιπέδων εκπομπών και τα επίπεδα ρήπανσης μετρούνταν βάσει κάποιων ε, κοινών προδιαγραφών στις μεταφορές συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων δίζελ, με κινητήρες δίζελ. Αυτά που έγιναν εδώ πρόσφατα δείχνουν ότι οι εκπομπές αυτές που καταγράφονταν κατά τη διάρκεια δοκιμών ε, φαίνονταν να ήταν πολύ χαμηλότερες από την πραγματικότητα. Συνεπώς, οι εκπομπές των κινητήρων αυτών είναι πολύ πιο ψηλές από ό,τι φαινόταν και γινόντουσαν αποδεκτές Τις διάφορες δηλώσεις σχετικά με οχήματα τέτοιων κινητήρων. Σε αστικές περιοχές το επίπεδο των εκπομπών από τις μεταφορές είναι πολύ υψηλό και είναι μεγάλο το ποσοστό στα πλαίσια των συνολικών ε, ρηπάνσεων και πολύ υψηλότερο μάλιστα από ό,τι είχε υπολογιστεί αρχικά από τις χώρες μέλη. Οπότε η ερώτησή μου είναι, οι χώρες μέλη δεν θα έχουν κάποια ευθύνη για να κάνουν κάτι παραπάνω, να αναλάβουν την ευθύνη των υψηλότερων εκπομπών που είχαν στην πραγματικότητα από ό,τι αρχικά υπολογισμένες. Συνεπώς, εδώ περνάμε σε, μια, σε ένα δεύτερο επίπεδο σκέψης που λέει ότι κάποιες κατηγορίες κινητήρων diesel τα αυτοκίνητα έχουν στην πραγματικότητα πολύ ψηλότερα επίπεδα ρήπανσης από αυτά τα οποία λάβαμε υπόψη μας στις ε, διάφορες ρυθμίσεις. Και όταν έχουμε προγράμματα εθνικά μείωση των εκπομπών, δεν θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη αυτή η διαφορά. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Άλλος, παρακαλώ. Ναι, μία ερώτηση πάνω σε αυτό. Γιατί αναφέρθηκε το RD, αλλά υπάρχει τεράστια συζήτηση και υπάρχει και θέμα ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της απόφασης που Θα μπορούσατε στην ανάλυση σας παρακαλώ να μας πείτε ότι αυτή η δείχτες ψηλής συμμόρφωσης που συζητιούνται το 2,1 και στη συνέχεια 1,5 του Συμβουλίου και τώρα στο κάς αλλάζουμε τις προδιαγραφές στο 120. Σύμφωνα με τη δικιά σας την ανάλυση λοιπόν, ποια θα είναι η συνέπεια των διαδικασιών όσον αφορά το οξύδια του αζότου στις διάφορες χώρες και για το 2020 και για το 2030. Τι συνέπειες θα έχουμε στην ποιότητα του αέρος. Θα ήθελα να ξέρω την ε, άποψη της Γενικής Διεύθυνσης ΕΝΔΗ για την απόφαση αυτή RDE με ιδιαίτερα υψηλού δείχτες συμμόρφωσης όσον αφορά την ποιότητα του αέρος. Άλλη ερώτηση? Όχι. Ωραία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν απαντήσει παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως έχει πει επανελειμμένως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για διάφορους στόχους. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ καλή προκειμένου να μειώσουμε την ρήπανση και τις εκπομπές. Πιστεύουμε ότι με τα σημερινά μέτρα θα έχουμε σημαντικές επιπτώσεις και στην ποιότητα του αέρος. Δεν έχω βέβαια τίποτα στοιχεία, ούτε τίποτα πιο συγκεκριμένο, αλλά οι χώρες μέλη πρέπει έτσι καλώς μέχρι το 2020 να έχουν τηρήσει τις τιμές για τις οποίες έχουν δεσμευτεί. υπάρχει η ανάγκη για να γίνει αυτό και αυτό συγχρόνως σημαίνει ότι οι εκπομπές των οχημάτων αυτών που όπως είπατε ήταν υψηλότερε πρέπει να αντισταθμιστούν με κάτι άλλο για να τηρηθούν ε, οι στόχοι σε εθνικό, περιφερειακό επίπεδο, με άλλα μέσα, ό,τι μέτρα και να είναι, οι χώρες μέλη πρέπει να σκεφτούν κάτι. Για το στόχο για το 2030 όμως, αυτό παίζει μικρότερο ρόλο. Δεν πιστεύουμε ότι μέχρι τότε οι επιπτώσεις αυτής της διαφοράς θα είναι αισθητές. 2030 που θα είναι η επόμενη στόχη μείωσης. Ευχαριστώ πολύ, λέει και ο Πρόεδρος. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Με την πρώτη ερώτηση της δεύτερης ομάδας, διαδικασίες ε, επί παραβάσεως από την κυρία Κάτριν Μπέρντερ και δίνω στο το λόγο στην Κομισιόν για να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνούμε νομίζω με την εκφραστή άποψη ότι πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την εφαρμογή της οδηγίας για την ποιότητα του αέρος στα κράτη-μέλη και αυτό χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που έχουμε στη διαδικασία μας και αυτό περιλαμβάνει και τις διαδικασίες επί παρεμβάσεις. Ήδη από το 2008 έχουν υπάρξει υποθέσεις για την ε, παραβίαση των ε, ορίων για το EM10 από το 2005 και που εφαρμόζεται η σχετική οδηγία υπήρξε μια σημαντική προσπάθεια από τη δική μας πλευρά γιατί αφορούσε τις αξιολογήσεις 17 κρατών μελών. Και αν δούμε λοιπόν ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος να αντιμετωπίσουμε αυτές τις διαδικασίες επί παραβιάση. Στην περίπτωση 80 η Αυστρία συμμορφώθηκε εγκαίρος και δεν χρειάστηκε να έλθει ενώπιον της, ε, του δικαστηρίου. Αλλά υπήρξαν τέσσερα κατημέρια τα οποία καταδικάστηκαν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γιατί δεν συμμορφώθηκαν με τις οριακές τιμές για το EM10. Η απόφαση του δικαστηρίου φυσικά επιβεβαίωσε μονάχα τις προηγούμενες ε, παραβιάσεις και δεν μπόρεσαμε έτσι να χρησιμοποιήσουμε τα διαρθρωτικά, τα δομικά μέσα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τα κάτι μέλη προ μια συνεχιζόμενη συμμόρφωση στο μέλλον και γι' αυτό η Κομισιόν τροποποίησε την δική της όχι μόνο για να αντιμετωπίσει την υπέρβαση των αριακών τιμών αλλά και την ανεπάρκεια ή έλλειψη μέτρων που αφορούσαν διάφορες πηγές ε, ε, μικροσωματιδίων PM10. Και ξεκινήσαμε λοιπόν, ε, για να ξεκινήσουμε και άλλες διαδικασίες, χρειαζόμαστε πιο πολύ χώρο, γιατί είναι ένα πολύ πλοκό θέμα και είναι ένα σημαντικό εγχείρημα και δεν πρέπει να υποτιμήσουμε τους ανθρώπινους πόρους και το χρόνο που χρειάζεται για να εξετάσουμε την κατάσταση σε εκατοντάδες περιοχές όπου υπάρχει παραβίαση των ορίων αυτών πρέπει να το κάνουμε για τα 17 κράτη-μέλη και υπάρχουν, υπάρχει ανάγκη να υπάρξει απόδειξη για την παραβίαση αυτή, για την υπέρβαση των ορίων σε όλες τις περιπτώσεις σχεδόν. Έχει προχωρήσει η διαδικασία. Το, η Κομισιόν έχει παραπέμψει τη Βουλγαρία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που είναι η πιο ακραία περίπτωση στο φως των προηγουμένων εμπειριών Πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει επικύρωση από το, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο της προσέγγισης της Κομισιόν, εάν συμβεί κάτι τέτοιο, η απόφαση αυτή θα ισχύει και στο μέλλον και θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε και τις προσπάθειές μας έναντι άλλων καθομελών, τα οποία μπορεί να χρειαστεί να έρθουν ενώπιον του δικαστηρίου. Όπως όμως υπεγράφει, όπως υπεγραμμίστη από το έντιμο μέλλον δεν αφορούσε μοναχα την υπέρβαση των κανόνων PM10. Μετά από την ε, έλευση των οριακών τιμών το 2010 αντιμετώπιστηκαν και άλλες παραβιάσεις με τον ίδιο πλήρη τρόπο εν ώψη της σοβαρότητας της κατάστασης στο ΕΒ Η περίπτωση αυτή αντιμετωπίστηκε με προτεραιότητα ενώ συνεχίζονται οι διαδικασίες εναντίον και των άλλων κρατών μελών. Η έρευνες έχουν γίνει ήδη στα άλλα κράτη-μέλη όπου έχουν αναφερθεί παραβιάσεις και υπερβάσεις αυτών των οριακών τιμών και αυτό θα αφορά και τα 17 κράτη-μέλη. Μεταξύ αυτών δύο, έχουν, δύο υποθέσεις έχουν κλείσει διότι υπήρξε συμμόρφωση αλλά υπάρχουν έξι περιπτώσεις που έχουν δώσει λαβή σε διαδικασίες επί παραβιάση. Έχουν γίνει, ε, έχει γίνει έκδοση ε, αιτιολογημένης γνώμης στις άλλες περίπτωσεις και περιμένουμε την απάντηση των κρατών μελών. Κύριε Μάρτεν. Ευχαριστώ. Νομίζω πως ε, δεν υπάρχει βουλευτή στο Κοινοβούλιο που να μην έχει, το έχει ζητηθεί από τους ε, ψηφοφόρους του το τι κάνουν, τι κάνουν κάθε, όταν ψηφίζεται κάποια νομοθεσία και δεν εφαρμόζεται. Η νομοθεσία τώρα αφορά στο 2008. Μιλάμε ακόμα για ανάληψη δράσης, ε, προχωράμε τη διαδικασία παρα, παραβάση. Είναι κάπως ενοχλητικά όλα αυτά. Νομίζω πως τα κράτη-μέλη τα οποία διαφεύγουν μη συμμόρφωση τις κυρώσεις ε, και λένε εντάξει θα πέρασει κανένας χρόνος μέχρι να φτάσει η επιστολή θα έχουμε δύο-τρία χρονάκια μέχρι να το εξετάσουμε και να εξεταστεί όλο ζήτημα. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω, εντάξει ακούω το θέμα των δυσκολιών που υπάρχουν με τους ανθρώπινους πόρους. Αλλά αν, επειδή η Κομισιόν είναι ναι, ο χωροφύλακας σε ό,τι φορά την ε, νομοθεσία, ίσως θα πρέπει να αποκτήσει τα μέσα για να μπορεί να ασκήσει την κατάλληλη αστυνόμευση. Χρειάζεται να είμαστε πιο αυστηροί και να βρούμε με άμεσα απέναντι σε όλους τους παραβαίνουν. Πρόκειται για την ποιότητα ζωής, ε, του αέρα. Αυτό λοιπόν η αργοκίνητη μηχανική, ε, μηχανή μας καταπιέζει πολύ και όχι μόνο εμάς και σας ερωτώ υπάρχει κάποιος τρόπος που να, να θεωρήσετε ότι η Κομισιόν μπορεί να επιταχύνει τις διαδικασίες αυτές. Θα υπάρχουν οι τριμερείς διάλογοι, συζητήσεις που διεξάγονται συνεχώς για να πετύχουμε μια τελική συμφωνία και μετά περνάνε καμιά δεκαετία χρόνια μέχρι ότου να επιτευχθεί η συμμόρφωση. Είναι πραγματικά δυσάρεστο και θλιβερό για όλους μας εμείς ε, οι βουλευτές που συναντάμε τους, ε, το εκλογικό μας σώμα και συνεχώς μας ερωτών διότι, γιατί δεν φροντίζεται να επιβληθεί η νομοθεσία την οποία έχετε ψηφίσει. Thank you. Ευχαριστώ. Ναι, όλοι μπορούν να κατανοήσουν ε, αυτή την απογοήτευση. Είναι μια διαδικασία που θα πρέπει να εξεταστεί τρόπο ουσιαστικό. Εδώ μιλάμε για 17 κράτη-μέλη, εκατοντάδες περιοχές που είναι υπερβάσεις ορίων και θα πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας με τέτοιο τρόπο ώστε να ε, επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα και να υπάρξει ιδέουσα επιμέλεια. Πρέπει να βάλουμε λοιπόν όλους τους πόρους για όλες τις προσπάθειες που έχουμε για να κερδίσουμε μια υπόθεση που έχει, έχει φτάσει στο δικαστήριο. Χρειάζεται νομική δουλειά και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο ε, αυτές οι διαδικασίες χρειάζονται πολύ χρόνο. Υπάρχουν και διαδικασίες ε, που δεν είναι στο χέρι μας να τις αλλάξουμε πρέπει να τις ακολουθήσουμε. Έχουν αποδειχθεί ότι είναι οι ορθές, οι σωστές, αλλά είναι γεγονός πως ε, το κοινό μπορεί να δυσαρεστείτε, Αλλά φυσικά δεν σταματάμε μόνο στη διακασία επί παραβάση. Και υπάρχει κάτι που έχει γίνει πιο σημαντικό στην πολιτική μας, δηλαδή όταν κρίνουμε πως ε, ένα κράτος μέλος ε, κινδυνεύει ή ήδη έχει υπερβεί τα σωριακές τιμές, τότε ερχόμαστε σε στενή επαφή με τον λόγο συζητάμε τουλάχιστον με του εκπροσώπους της, ε, των περιοχών, των πόλεων, για το τι πρέπει να γίνει. Έχουμε λοιπόν μια παράλληλη διαδικασία η οποία προχωράει και προσπαθούμε να πετύχουμε να μην υπάρξουν πλέον υπερβάσεις και να κλείσουμε με την διαδικασία επί παραβάση. Αλλά το πιο σημαντικό είναι οι υπερβάσεις ε, να πάψουν να υφίστανται και, τα, και οι πολίτες να έχουν την ε, διασφάλιση ότι ο αέρας που αναπνέουν είναι καθαρός. Αυτά τα παράλληλα μονοπάτια θα έλεγα που να τα εφαρμόσουμε τα τελευταία χρόνια. Κάποια κράτη-μέλη έχουν συμμορφωθεί και πιστεύουμε ότι και άλλα κράτη-μέλη θα ακολουθήσουν αυτήν την άγουσα. Επιταχύνουμε ε, το, το δυνατόν αυτές τις διαδικασίες μέσω αυτών των παράλληλων οδών που ακολουθούμε. Ευχαριστώ. Πολύ. Τώρα, έκθεση στο σωματίδιο. Έχουμε εδώ και την κυρία Πέρντε. Ποιος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Λέει η Επιτροπή. Όπως είπα και πριν, υπάρχουν πολλές χώρες που ξεπερνούν τα όρια. Πολλές βλέπουμε ότι αυτοί που επηρεάζονται μειώνονται σε αριθμό. Τα προβλήματα έχουν κυρίως να κάνουν με την σετήσιες και τις ημερήσιες τιμές. Θα πρέπει να έχουμε ή το ένα ή το άλλο. τουλάχιστον να υπάρχει συμμόρφωση με τις αιτήσιες τιμές. Είναι σοβαρό το ζήτημα σε κάποιες χώρες μέλη, είναι αλήθεια. Η εμπειρία όμως από άλλες δείχνει ότι υπάρχει συμμόρφωση πολλές φορές και άρα υπάρχουν ελπίδες. Οι προβολές που κάναμε δείχνουν ότι στις περισσότερες χώρες μέχρι το 2006 το πολύ θα πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση από όλες τις χώρες μέλη. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει δράση. Πρώτον, κατά της Βουλγαρίας, γιατί εκεί υπάρχει διαφορά και ο κίνδυνος στον πληθυσμό είναι πιο μεγάλος, αλλά παρακολουθούμε από κοντά την κατάσταση και στις υπόλοιπες χώρες μέλη. Έχουμε ήδη επιπλέον αιτιολογημένη γνώμη και ίσως ακολουθήσει και άλλη δράση ανάλογα με το τι θα δούμε. Αν δούμε ότι οι χώρες ε, μέλη έχουν ή δεν έχουν συμμορφωθεί. Οι στόχοι περιβαλλοντικοί που αναφέρονται στην οδηγία έχουν νομικό καθεστώς όσον αφορά την εφαρμογή τους για το PM10 είναι σαφές, είναι σαφής υποχρέωση, αλλά για άλλα στοιχεία έχουμε την τιμή στόχο. που επιτρέπει περισσότερη ευελιξία στις χώρες μέλη. Ανάλογα και με την φύση της κατάστασης στην αλυσίδα του όσοντος. Η έγκριση της νέας οδηγίας έχει μεγάλη σημασία. Πολλές φορές διαπιστώνουμε τα προβλήματα στην αλυσίδα του όζοντος σε άλλες χώρες από εκείνες που έχουμε τις υψηλές εκπομπές. Οι χώρες μέλη μπορούν να είναι σίγουρες ότι μπορούν να πετύχουν τη μείωση των εκπομπών τους και άρα να τηρήσουν τις οριακές τιμές όσον αφορά τη ρήπαση της ατμόσφαιρας. Ευχαριστώ. Κυρία Μπέρδερ. συνδέεται με το προηγούμενο ερώτημα, δηλαδή πώς μπορεί κανείς να λειτουργήσει με γρήγορο ρυθμό με τις χώρες αυτές και φυσικά εδώ έχουμε μια κατάσταση όπου τα πράγματα έχουν γίνει πιο περιφερικοποιημένα. Μια νομοθεσία θα πρέπει να καλύπτει όλους τους τομείς μιας οικονομίας οι οποίοι θα συμμετέχουν. Πρέπει όλοι οι τομείς λοιπόν να συμβάλλουν. Ελπίζουμε λοιπόν ότι αν συνεργαστούν όλοι οι τομείς θα είναι πιο εύκολο να δώσουμε μια λύση για τα θέματα αυτά. Αλλά όταν έχουμε 20 κάτι μέλη τα οποία δεν συμμορφώνται και συμμορφώνται μόνο τα 8, τι θα λένε. Αν όλα τα άλλα κράτη δεν συμμορφώνται, πώς θα πείσετε ένα κράτος να κάνει κάτι. Και αν ε, εστιάζεται μονάχα σε ένα κράτος μέρος όπου η κατάσταση είναι ιδιαίτερα οξία Πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά τα θέματα για την Κομισιόν. Πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε την νομοθεσία όταν έχουμε να κάνουμε τέτοιες καταστάσεις. Κατανοώ αυτά που λέτε, αλλά νιώθω μια ματέωση. Πάρα πολλοί καταφέρνουν να έχουν υψηλή ρήπανση και ξεφεύγουν ουσιαστικά από τις κυρώσεις και δεν βλέπουμε ότι το αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό αποτελεσματικά. Δεν προστατεύουμε την υγεία του κόσμου αν ήταν δηλητηριασμένο νερό βέβαια το οποίο έβγαινε από, τα, από τις βρύσες, ναι θα κάναμε κάτι περισσότερο, είναι πιο εύκολο από την περίπτωση του αέρα. Αλλά αυτό είναι κάτι όπου λέμε ναι, βγάζουμε δείγματα εδώ, βγάζουμε δείγματα εκεί, αλλά δεν πάμε πουθενά. Σας ευχαριστώ παρόλα αυτά για την απάντησή σας. Καταλαβαίνετε, δεν είναι το πιο απλό θέμα. Και νομίζω ότι το θέμα της μη συμμόρφωσης αρχίζει να γίνεται όλο και πιο έντονο στην, ε, στα μάτια της κοινή γνώμης. Ευχαριστώ. Λέει Είναι 16, όχι 20 τα κράτη τα οποία δεν συμμορφώνονται και δεν είναι το σύνολο κάθε κράτους μέλους. Νομίζω ότι εδώ χρειάζεται μια σαφήνεια πολλές φορές είναι ορισμένα συγκεκριμένα σημεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για αυτούς που ζουν εκεί, αλλά δεν μιλάμε για ολόκληρες επικράτειες ενός κράτους, το σύνολο της επικράτειας ενός κράτους μέλους. Και αντιμετωπίζουμε το θέμα των παραβιάσεων σταδιακά και γιατί πιστεύουμε ότι καλύτερα να ξεκινήσουμε εκεί που το πρόβλημα είναι το πιο μεγάλο και που υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος για τον πληθυσμό ο οποίος εκτίθεται εκεί. Αλλά θέλω να το τονίσω και πάλι, παρακολουθούμε όλες τις περιπτώσεις όπου υπάρχει υπέρβαση των ορίων, αλλά φυσικά οι προτεραιότητές μας θα πρέπει να θεσπίζονται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, θα πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα με τα πιο σοβαρά προβλήματα, χωρίς αυτό να σημαίνει παραγνωρίζουμε τις άλλες παραβιάσεις τα βλέπουμε τα πράγματα συνολικά. Thank you Ευχαριστώ. Έκτη ερώτηση. Στις περιοχές του Λεγκρέσιου και του Άγου Βερσάνο και αυτό αφού είναι η ερώτηση του κ. Πετιτσίνη. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Πολλά στοιχεία υπάρχουν εδώ. Αρχίζω με την ποιότητα του αέρος. Ίσως επαναλαμβάνομαι εδώ, αλλά πρέπει για να είναι σαφές. Αξιολογούμε την αποδεχτή από τις χώρες μέλη ποιότητα του αέρος ετησίως. Για το 2014, για παράδειγμα, τα περιμέναμε για το Σεπτέμβριο. Προς το παρόν έχουμε διαδικασίες κατά ε, παραβάση κατά της Ιταλίας που συμπεριλαμβάνει και τη 1501 και το Ριζαναμέντο Νάπολη και Κασέρτα. καλύπτει δηλαδή η διαδικασία αυτή επί παραβάση, αυτή την περιοχή ακριβώς. Όσον αφορά το είδωρ, υπενθυμίζουμε ότι οι χώρες μέλη έχουν την υποχρέωση να ερευνούν και να διορθώνουν την κατάσταση όσον αφορά τις ε, προδιαγραφές για το ίδιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει πώς εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές οι χώρες μέλη και πρόσφατα έχουμε συστήσει για την Ιταλία, ειδικά και γενικά μέτρα για να αντιμετωπιστεί η ρήπανση από χημικά σε περιοχές κοντά σε εργοστάσια και η χώρα μέλος μέσα στο 2015 θα έπρεπε να εγκρίνει σχετικά μέτρα έτσι, και θα τα υποβάλει το Μάρτιο του 2016 στην Επιτροπή μας. Υπενθυμίζουμε επίση ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει ήδη καταδικάσει την Ιταλία επειδή δεν συμμορφώθηκε με την οδηγία στον αφορά τα απόβλητα στην Καμπανία και επειδή δεν υπάρχουν και τα κατάλληλα δίκτυα ε, απομάκρυνσης αποβλήτων. Οι βιομηχανικές εκπομπές είναι νόμος και οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους τα μέτρα για να αντιμετωπιστεί η ρήπανση αυτή. Τώρα, αν πρόκειται για κάποια παραβίαση, είτε για τον αέρα, είτε για το είδωρ, τότε η αρμόδια εθνική αρχή μπορεί να προτείνει επιπλέον μέτρα και να τα εφαρμόσει. Και αν υπάρχει παράβαση, οι αρχές μπορούν να πάρουν μέτρα για να επιβληθεί συμμόρφωση. Δεν έχουμε συγκεκριμένη πληροφορία για κάποια μονάδα βιομηχανική στο Βάλλοντο Λίτσιο Λεγκρέο στην Καμπανία αλλά για άλλες μονάδες που αναφέρονται στις μελέτες. Πρέπει να πούμε ότι έχουμε ξεκινήσει κατά της Ιταλίας διαδικασία επί παραβάση εξαιτίας της ρήπανσης από μία βιομηχανική ομάδα, ε, μονάδα. Συνεπώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δραστηριοποιείται προκειμένου να διορθωθούν όλα αυτά τα ζητήματα για τα οποία κρίναμε ότι υπάρχει παραβίαση της κοινοτική περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την κυρία Διευθύντρια για την απάντησή σας. Από ό,τι θυμάμαι βρισκόσασταν σε μια εκδήλωση που μιλήσαμε για το Τέραντι και ακούσαμε τι φωνές απόγνωσης αυτών των ε, κατοίκων. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με το αποστάσιο της Ήλβα στον Τάραντο. Ε, κατά την άποψή μας ε, εδώ χρειάζεται μια πιο στεναρή παρέμβαση. Μια παρέμβαση πιο στεναρή ε, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιπαραβάση. Πιστεύω πως απαιτείται μια πραγματική παρακολούθηση της διαχείρισης ε, του προβλήματος από πλευράς ε, Ευρώπης και Κομισιόν και όχι μια τοπική διαχείριση των πόρων που ε, χρησιμοποιούνται για την εξυγίανση διότι σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι ιδιαίτερα διεφθαρμένο θα πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζεται αυτή η πόσο έλεγχο Η Ευρώπη δικάνει, δίνει νέου πόρου και το σύστημα διατηρεί αυτήν την κρισιμότητα της κατάστασης εις βάρος των πολιτών. Δεν αρκεί λοιπόν η προσφυγή παραβάση. Γι' αυτό είχα ζητήσει την Επιτροπή Περιβάλλοντος να μεταβεί στον Τάραντο, δεν ξέρω πότε θα πάμε, αλλά είναι σημαντικό να πάμε για να δούμε με τα ίδια μας τα μάτια το τι συμβαίνει δεν θα επιληθεί το ζήτημα αγαπητή Διευθύντρια μέχρι το, μέχρι το Μάρτιο 2016 εάν όλοι δούμε με τα μάτια μας αυτά που είδα εγώ. Εάν κατανοήσουμε και συνειδητοποιήσουμε ότι πρόκειται για μια καταστροφική περίπτωση όπου η διαδικασία παραβάση δεν θα αρκέσει. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν θέλει να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Επόμενο θέμα είναι η αναθεώρηση των τρεχουσών διατάξεων. Έχουμε την κυρία Βέροντολ για την ερώτηση παριθμών 7. Και θα δώσω το λόγο στην Κομισιόν για να απαντήσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι έχει καταστεί σαφές πως ε, η οδηγία είναι ένα θέμα κλειδί. Αν θέλουμε να διασφαλίσουμε μελλοντικέ ε, συγκεντρώσει χαμηλότερες από αυτές του ΠΟΗ και να το διασφαλίσουμε πανταχού. Το 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια ε, επισκόπηση της ευρωπαϊκής πολιτικής και αυτή η επισκόπηση κατέδειξε ότι δεν είναι κατάλληλο να ε, υπάρξει αναθεώρηση της συγκεκριμένη ε, οδηγίας. Να υπενθυμίσω ότι οι οριακές τιμές συμπίπτουν με αυτές του ΠΟΗ για πολλούς ρηπαντές και βρήκαμε και κάποιες βασικές αποκλήσεις ε, στα όρια που υπάρχουν και για το PM10 και για το PM2,5. Για το PM10 ξέρετε ότι 60 κρατημένοι ε, μίλησαν για ε, υπέρβαση ακόμα και με τα λιγότερο αυστηρά όρια της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι ε, θα χρειάζεται να πετύχουμε τη συμμόρφωση με τις ωριακές ε, τιμές για το PM2,5 εφαρμόζονται από τον Ιανουάριο ανεστώτος έτος θα πρέπει να λάβουμε τις απαραίτητες προφορίες για να αποκτήσουμε μια γενικότερη εικόνα σχετικά με την συμμόρφωση. Το πρόγραμμα της Κομισιόν για καθαρό αένα το οποίο ξεκίνησε το 2013 εστιάζει στην επίτευξη συμμόρφωση με τα εφιστάμενα όρια μέχρι το 2020 και χρησιμοποιώντας μια αναθεωρημένη οδηγία NEC για την ε, ρήπανση για αυτές οι μειώσεις ε, σίγουρα θα πρέπει να ισχύσουν για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η, η οδηγία περί ποιότητας του αέρα θα πρέπει να ε, βρίσκονται σε στενή παρακολούθηση, να λαμβάνουμε υπόψη όλε τις προφορίε, ειδικά για το VM2,5, για το μονοξίδιο του αζότου και θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτέ τι ευκαιρίες, αυτέ τι επισκοπήσεις ε, όταν θα είναι διαθέσιμε σε κάνα δύο χρόνια και προς το παρόν χρειάζεται να διασφαλίσουμε πως όλα τα κρατημέλη εφαρμόζουν τα και τηρούν τα όρια προτού να λάβουμε νέα μέτρα για να ευθυγραμμιστούμε με τις κατηγραμμές του ΠΟΗ. Δεν ξέρω αν θέλετε ε, ναι, εδώ μοιραζόμαστε τη δουλειά, λέει ο κύριος ε, Ερμπράντη. Σας ευχαριστώ κυρία μου για την απάντηση της ε, ερώτησης εκ μέρους της Κομισιόν. Κατανοώ τη δυσκολία που έχει η Κομισιόν να καταλήξει σε μια απόφαση γιατί γνωρίζει ότι για επιστημονικούς λόγους ότι είναι απαραίτητα πιο αυστηρά πρότυπα, αλλά συγχρόνως έχει να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα στα κράτη-μέλη που <clears throat> δεν συμμορφώνται ούτε καν με τους τωρινούς κανόνες, πόσο μάλλον με μελλοντικού αυστηρότερους κανόνες. Είναι παράξενο όμως ότι εμείς ουσιαστικά ανταμείβουμε τα κράτη-μέλη για την παραβίαση των τωρινών προτύπων γιατί αυτό σημαίνει ότι αυτοπεριοριζόμαστε σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε πιο ψηλά επίπεδα προστασίας ακολουθώντας αυτά που ζητά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Το ερώτημα μου προς την Κομισιόν είναι το εξής. Εγώ κατανοώ για την νομοθεσία ότι πολιτικά δεν είναι εφικτό να προτείνει κανείς πιο αυστηρά πρότυπα για την ποιότητα της, ε, του, αέρα. Αλλά σε επικοινωνία με τα κράτη-μέλη. Φαντάζομαι ότι η Κομισιόν αναφέρεται πάντα στις κατευθυντές γραμμές του ΠΟΕ για να του, του ΠΟΗ, του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, για να καταλάβουν τα κράτη-μέλη ότι δεν φτάνουν οι τωρινοί κανόνες, αλλά σε ένα ιδανικό κόσμο θα έπρεπε να έχουν ακόμα πιο ψηλά πρότυπα. Είναι κάτι το οποίο το αναφέρεται συνέχεια από την Κομισιόν προς τα κράτη-μέλη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Βεβαίω, απολύτως, πλήρω. Όταν είπα προηγουμένως ότι είμαστε σε επαφή με τα κάτι μέλη σε σχέση με τα θέματα αυτά, όχι μόνο για τι επί παραβάσει διαδικασίες, μιλάμε και με τοπικές αρχές, με τις πόλεις, όχι μόνο με την κεντρική κυβέρνηση. Πάντα τονίζουμε ότι στο μέλλον θέλουμε να φτάσουμε να εφαρμόσουμε τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και αυτό είναι κάτι το οποίο το είπαμε όταν ε, παρουσιάσαμε τις ε, αναθεωρημένες οδηγίες ΝΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Και ξέρουν όλοι ότι οι προτάσεις μας θα πρέπει να ε, μειώσουμε τον αντίκτυπο της ρήπανσης του αέρα και να πλησιάσουμε πιο κοντά στις κατευθυντήρες γραμμές του ΠΟΕ. Από τη στιγμή τώρα που όλα αυτά έχουν τεθεί εν κίνηση και βλέπουμε ότι και οι κανόνες του ΠΟΗ για ορισμένε ρηπαντικές ουσίες είναι υπό αναθεώρηση, μπορούμε να πούμε ναι, θα παρακολουθήσουμε όλα αυτά τα στοιχεία και θα πάρουμε τις δικές μας αποφάσεις για το αν υπάρχει, αν χωρεί ανάγκη να πράξουμε κάτι και αν είναι αυτό απαραίτητο να αναθεωρήσουμε τις οριακές τιμές. Αν δείτε την ποιότητα του, της ατμόσφαιρας στην Ευρώπη μετά από την έκθεση που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, βλέπετε είναι στοιχεία και υπάρχει φρασιολογία που είναι πολύ σαφής λέει ότι τελικά πρέπει να φτάσουμε τους στόχους του ΠΟΗ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ζητώ από την Κομισιόν να μας πει αν μπορεί να απαντήσει τι τις δύο τελευταίες ερωτήσεις που έχουν τεθεί Η ερωτούσα βρίσκεται σε μια άλλη συνεδρίαση του Κοινοβουλίου. Έχουμε την ερώτηση παρέθμων 3 για την παραβίαση ετησίων ορίων καθώς και την ερώτηση 8 για, μάλλον γιατί τις ερωτήσεις 3 και 8 που αφορούν και οι δύο την παραβίαση σε σχέση με τα οξύδια του αζώτα από τα αυτοκίνητα της. μπορεί να απαντήσει η Κομίσιο, βέβαια, μπορώ για το ερώτημα υπαριθμών 3. Μετά από την έρευνα που έγινε για όλα τα κράτη-μέλη που έχουν ε, αναφέρει υπερβάσεις των ε, ορίων για το διοξίδιο του αζότου, έχουμε ξεκινήσει διαδικασίες που αφορούν τις πιο σοβαρές περιπτώσεις επί τη βάση των δύο κριτήριων που αναφέραμε προηγουμένως, το ύψος της υπέρβασης και το μέγεθος του εκτεθειμένου πληθυσμού. Βάσει των πληροφοριών των κρατών μελών αξιολογούμε την κατάσταση. Στην επόμενη χρονική διά, ε, διάρκεια, στο επόμενο χρονικό διάστημα, θα έχουμε ένα δεύτερο κύμα διαδικασιών που μπορεί να κινηθούν εναντίον άλλων κρατών μελών και φυσικά οι τωρινές διαδικασίες επί παραβάση μπορεί να αναβαθμιστούν <clears throat> αν δούμε ότι δεν γίνονται οι απαραίτητες εθνικές ενέργειες για να αντιμετωπιστούν τα θέματα αυτά, θα προχωρήσουμε περαιτέρω. Αυτό ήταν για το ερώτημα 3. Για το ερώτημα είπα αριθμόν 7. 8 καλύτερα. Για τα όρια διοξιδίου του αζότου από τα αυτοκίνητα δίζελ το έχουμε αναφέρει το θέμα αυτό και σας είπα ότι η Κομισιόν έχει δράσει με μεγάλη αποφασιστικότητα για να εξασφαλίσει την αξιοπιστία του νομικού συστήματος, του δικαστικού συστήματος, να εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, αλλά πάνω απ' όλα για να μην υπάρξει πρόσφατη ε, βλάβη στην ε, υγεία των πολιτών και το περιβάλλον μας και για να εξασφαλίσουμε ότι οι δοκιμασίες των οχημάτων θα γίνουν με τρόπο ανθεκτικό και που εξασφαλίζουν την αξιοπιστία τους και ξέρουμε ότι από το 2020 θα τροποποιηθεί η τεχνολογία η οποία χρησιμοποιείται και όσο βελτιώνεται αυτή η τεχνολογία θα μειωθεί το περιθώριο σφάλματος. Όπως αναφέρθηκε και στο θέμα των πραγματικών τεστ για τις εκπομπές, αυτό είναι μόνο μια μια πτυχή του προβλήματος πρέπει να εξετάσουμε καλύτερα τα θέματα της έγκρισης τύπου και της παρακολούθησης της ε, αγοράς και η Κομισιόν εργάζεται ήδη από τη βάση προτάσεων για να κάνει πιο στεναρή και ανθεκτική την διαδικασία έγκρισης τύπου και να δημιουργήσει μια εργαλειοθήκη για να μπορέσει να αναλυφθεί δράση για προϊόντα τα οποία δεν είναι ασφαλή εστίαση εδώ είναι να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τη διασφάλιση των διαδικασιών και να υπάρξει κατάλληλη συνεργασία μεταξύ των αρχών που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή αυτού του νομοθετήματος και επίσης τα κράτη-μέλη θα υποχρεωθούν να προχωρήσουν σε παρακολούθηση της αγοράς και να κάνουν ελέγχους στα αυτοκίνητα που μπαίνουν στην αγορά <clears throat> και τέλος θα υπάρξει μεγαλύτερη δυνατότητα της Κομισιόν να παρεμβάνει και να αποφασίζει για τις διορθωτικές δράσεις των κρατών μέλων. Και αυτά τα μέτρα θα περιληφθούν σε ένα σχέδιο πρότασης για τη μεταρρύθμιση του Γενικού Πλαισίου Έγκρισης Τύπου που σύντομα θα εγκριθεί. διαμέσως παρακολουθούμε προσεκτικά τις ε, απόψεις που έχουν εκφραστεί για άλλες δυνητικές δράσεις μεταξύ των οποίων και η ανάγκη να υπάρξει ένα αποτελεσματικό σύστημα εποπτείας και παρακολούθησης ή ένας ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης. Και είμαστε έτοιμοι να διερευνήσουμε όλες αυτές τις δυνατότητες υπό την έποψη του κόστους και της εφικτότητας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Άλλος κανείς. Όχι από ό,τι βλέπω. Ευχαριστούμε πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εδώ τελειώνει η συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Ένδυ. Η επόμενη συνεδρίασή μας είναι στις 14 στις 3 Δεκεμβρίου έχουμε την κοινή με την ε, Άγκρη και μετά στις 14 Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο. Ευχαριστώ πολύ.